So, good afternoon. Καλό απόγευμα σε όλους. Θα ήθελα να καλωσορίσω εδώ σήμερα τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο, τον κύριο Τομπρόφσκι και το, τους επιτρόπους Τζεντιλόνι και Σμιτ για οικονομικό διάλογο πάνω στην φθινοπορεινή δέσμη μέτρων ε, πάνω στο ε, Ευρωπαϊκό Εξάμεινο 2020. Η δέσμη αυτή ξεκινάει τον κύκλο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με συστάσεις για την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ ε, την ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη, ε, το, την ε, έκθεση για, και την κοινή έκθεση απασχόλησης. Ο σημερινός διάλογος αποτελεί τμήμα του πλαισίου που συμπεριλαμβάνεται στη δέσμη 6 μέτρων. Πιο συγκεκριμένα, ο διάλογος αυτός επιτρέπει στους συγητές και σκιώδεις συζητητές των εκθέσεων πρωτοβουλίας για την ετήσια επισκόπηση ανάπτυξης και την κοινή έκθεση απασχόλησης να συμμετάσχουν σε ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα δώσω τώρα το λόγο στους επιτρόπους ε, για να μας ε, παρουσιάσουν τις αρχικές τους ε, παρατηρήσεις. Έξι λεπτά στον καθένα. Κύριε Τομπρόφσκης. Κυρία Πρόεδρε, ε, κύριοι Ευρωβουλευτές, ε, συνάδελφοι, χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ για την πρώτη ανταλλαγή απόψεων πάνω στην ε, δέσμη μέτρων για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας. Πάντα εκτιμούσα την συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία του εξαμήνου, διότι μας παρουσιάζεται ενδιαφέρουσες προοπτικές. Οι συζητήσεις μας πάντα ήταν ανοιχτές και επίκαιρες. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή όσον αφορά το ευρύτερο οικονομικό πλαίσιο. Η ευρωπαϊκή οικονομία ε, βρίσκεται τώρα στην 8η ε, ε, χρονιά ανάπτυξή τη. Η απασχόληση βρίσκεται σε επίπεδα ρεκόρ, οι επενδύσει αυξάνονται και έχουν βελτιωθεί, έχει βελτιωθεί η δημοσιονομική κατάσταση. Ωστόσο υπάρχουν κάποιε αποκλήσει με υψηλή ανεργία σε κάποια κράτη-μέλη και επίση αντιμετωπίζουμε κινδύνους που σχετίζονται με τι εξωτερικέ προοπτικέ και τι γεωπολιτικέ εντάσει. Επιπλέον αναμένονται σημαντικές αλλαγές στις επόμενες επόμενε δεκαετίε, συμπεριλαμβανομένη τη αλλαγή του κλίματο ε, και τη ε, μετάβαση ε, σε μια οικονομία με χαμηλέ εκπομπέ οξυδιού του άνθρακα, τεχνολογικέ αλλαγέ, ψηφιοποίηση και τιμογραφική αλλαγή, οι οποίε θα μεταμορφώσουν θεμελιωδώ τι οικονομίε και κοινωνίε μα. Θα πρέπει να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί με τρόπο βιώσιμο και δίκαιο. Η ετήσια στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης ε, θέτει τις ε, οικονομικές ε, και προτεραιότητες για την Ευρωπαϊκή Ένωση και επικεντρώνεται στην ανταγωνιστική βιωσιμότητα. Ε, η αυτή η ονομασία αντικατοπτρίζει ε, ε, ένα βιώσιμο και συμμετοχικό οικονομικό μοντέλο που βασίζεται σε τέσσερι αρχέ: σταθερότητα, παραγωγικότητα, δικαιοσύνη και βιωσιμότητα. Καταρχά, η οικονομική σταθερότητα αποτελεί προπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη. Χρειάζεται οι δημοσιονομικέ πολιτικέ να είναι υπεύθυνε και διαφοροποιημένε, ώστε να έχουμε βιώσιμη δημοσιονομική κατάσταση σύμφωνα με του συμφωνηθέντε κανόνε. Τα κάτι μελη με ε, δημοσιονομικό περιθώριο θα πρέπει να το εκμεταλλευτούν ενώ η μείωση του χρέους ε, είναι κάτι που οδηγεί σε ε, περισσότερη αυτοπεποίθηση. Ε, και καλύτερη αντοχή για τις χώρες αυτές. Επιπλέον ε, θα πρέπει να ε, ελεγχθούν οι ανισορροπίες που υπάρχουν και ο Πάολο θα αναφερθεί περαιτέρω στο θέμα αυτό. Ταυτόχρονα χρειάζεται επίσης να προωθήσουμε τις εργασίες μας πάνω στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και της Ένωσης Κεφαλογορών είναι απαραίτητε για να έχουμε ισχυρή Ευρώπη στην διεθνή σκηνή. Δεύτερον, παραγωγικότητα. Ε, ο πληθυσμός ε, γυράσκει και ε, έχουμε όλο και πιο περιορισμένους πόρους και γι' αυτό η ανάπτυξη εξαρτάται από την υψηλή παραγωγικότητα και την καινοτομία. Επενδύσεις στην εκπαίδευση, διαρθρωτικές αλλαγές θα πρέπει να επιτρέψουν τις επιχειρήσεις να ωφεληθούν από τις καινοτομίες, προωθώντας έτσι την παραγωγικότητα. Χρειαζόμαστε ανταγωνιστικές και αποτελεσματικές αγορές. Τρίτον, δικαιοσύνη. Η κοινωνική δικαιοσύνη βρίσκεται στον πυρήνα του, της ε, ευρωπαϊκής οικονομίας ε, και στην, ε, στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εσείς και το Συμβούλιο έχουν τονίσει τη σημασία του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ε, και ε, είμαστε προσιλωμένοι στην ε, εφαρμογή του. Επίσης, θα πρέπει να φροντίσουμε η νέα ψηφιακή οικονομία να είναι δίκαιη. Μόλι έχουμε δημοσιεύσει μια ανακοίνωση που λέγεται «Ισχυρή κοινωνική Ευρώπη και δίκαιη μετάβαση». Η φθινοπορεινή δέσμη μέτρων προβλέπει ε, και ε, μάλλον παρουσιάζει τις βασικές εξελίξεις ε, στην απασχόληση και τον κοινωνικό τομέα. Η ανάλυση μας επιβεβαιώνει ότι η Ευρώπη κάνει πρόοδους όσον αφορά την εφαρμογή του πυλώνα. Ε, και ε, θα αναφερθεί περαιτέρω Νικολά στο θέμα τη ε, σύγκληση. Η τέταρτη αρχή είναι η βιωσιμότητα. Η Ευρώπη θα πρέπει να γίνει η πρώτη ήπειρο που να είναι ουδέτερη ω προς το κλίμα και αυτό αποτελεί πρόκληση για την γενιά μα. Η αλλαγή του κλίματο δεν σταματάει στα σύνορα και επηρεάζει όλου μα. Η μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα θα απαιτήσει σημαντικέ επενδύσει. για να πετύχουμε τους ισχύοντες στόχους για το 2030 όσον αφορά το κλίμα και την ενέργεια ε, θα απαιτήσει 260 δισεκατομμύρια επιπλέον ε, επενδύσεων κάθε χρόνο. Γι' αυτό θα πρέπει να καταβάλουμε σημαντικέ προσπάθειε σε όλα τα επίπεδα, ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό. Ε, δεν αρκεί μόνο ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει και τα κράτη-μέλη και οι ιδιωτικοί φορεί να ε, συμβάλλουν. Για να πετύχουμε αυτή, αυτό το στόχο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει ε, το, την Πράσινη Συμφωνία και το σχετικό επενδυτικό σχέδιο. Έτσι στέλνουμε σαφές μήνυμα στις δημόσιες αρχές, ε, τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές ότι θα πρέπει όλοι να σκεφτούμε με οικολογικό προσανατολισμό. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Το σχέδιο αυτό βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Καταρχήν σε χρηματοδότηση. Θέλουμε να κινητοποιήσουμε πόρους τουλάχιστον ενός τρισεκατομμυρίου για βιώσιμες επενδύσεις σε επόμενη δεκαετία. Δεύτερον, χρειαζόμαστε τις ε, σωστές ε, ε, συνθήκες για να έχουμε βιώσιμες επενδύσεις. Είναι, είναι σημαντική ανάγκη για σαφείς κανόνες. Και τέλος, χρειαζόμαστε και καλά προγράμματα, δεν αρκούν μόνο τα χρήματα. Θα παράσχουμε λοιπόν ε, την απαραίτητη εμπειρογνωσία. Θα ήθελα να κλείσω ε, λέγοντα ότι πιστεύω ότι έτσι ανταποκρινόμαστε στα ε, καλέσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ήταν κυρίω δύναμη όσον αφορά την προσπάθεια για μια οικονομία ουδέτερη ω προ εκπομπέ του διοξιδίου του άνθρακα. Τέλη Φεβρουαρίου θα έχουμε τις εκθέσεις αναχώρα και πρώτα θα ξεκινήσουμε με την ενσωμάτωση των στόχων βιώσιμη ανάπτυξη στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Ο Παύλο θα αναφερθεί περαιτέρω πάνω σε αυτό. Δεύτερον, ε, θα ε, ε, διατηρήσουμε τη μακροοικονομική και κοινωνική μα προσήλωση για να αντιμετωπίσουμε τι προκλήσει μα. Και τέλο, θα διαπιστώσουμε ποιε είναι οι περιοχέ που επηρεάζονται περισσότερο από την μετάβαση σε κλιματική ουδετερότητα και αυτό θα αποτελέσει τη βάση για τον διάλογό μα με τα κράτη-μέλη. Ε, για την κατάρτιση των σχεδίων ε, δίκαιη μετάβαση ανά περιοχή. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και προσβλέπω στη συνεργασία μαζί σα. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ κύριε Ντομπρόφσκη. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Παύλο Τζεντιλόνι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι μεγάλη χαρά για μένα που βρίσκομαι σήμερα εδώ ενώπιον των δύο κοινοβουλευτικών σας επιτροπών. Θα επικεντρωθώ σε τρία ζητήματα. Το ένα για το εξάμεινο και τις συστάσεις ε, για την Ευρωζώνη και επίσης θα αναφερθώ και στην έκθεση που αφορά το μηχανισμό επαγρύπνησης. Όπως ακούσαμε μόλις, εργαζόμαστε προκειμένου να συμπεριλάβουμε τους στόχους του ΟΗΕ για την βιώσιμη ανάπτυξη στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Ξεκινήσαμε τη διαδικασία αυτή ήδη με την στρατηγική μας για την ετήσια βιώσιμη ανάπτυξη. Την ετήσια μας στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη μάλλον που σας παρουσιάστηκε. Ο επόμενος γύρος θα είναι οι εκθέσεις αναχώρα που θα δημοσιοποιηθούν τέλος Φεβρουαρίου και θα χτίσουμε πάνω σε αυτήν τη νέα στρατηγική ανάπτυξης, εμβαθύνοντας περισσότερο σε θέματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, σε θέματα που έχουν να κάνουν με τις συνέργειες, τις αντισταθμίσεις ανάμεσα στο περιβάλλον, τα κοινωνικά και την οικονομική μας πολιτική. Επίσης, έχουμε και τα παρατήματα τα οποία αναφέρονται στις επιδόσεις των χωρών μελών σε κάθε έναν από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Η κάθε χώρα θα πρέπει να παρουσιάσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στα εθνικά ε, προγράμματα μεταρρυθμίσεων, κάτι το οποίο αναμένουμε για τον Απρίλιο. Και το έργο αυτό θα ληφθεί υπόψη στις δικές μας αναχώρα τάσει που θα είναι έτοιμες στα τέλη του Μαΐου. Αυτά τα οποία σας παρουσιάζω και αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο είναι ότι βρισκόμαστε στα πρώτα βήματα για το τι μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι ένας πειραματικός κύκλος όσον αφορά την ενσωμάτωση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ στην ε, δικιά μας Πράσινη Συμφωνία. Έρχομαι τώρα τις ε, συστάσεις όσον αφορά την Ευρωζώνη και τις διαφεροποίησεις που υπάρχουν. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε την Ευρωζώνη σαν να πρόκειται πραγματικά για 19 ξεχωριστές οικονομίες. Πρέπει να την βλέπουμε σαν μία οικονομική οντότητα. Και τα θετικά τα αποθέματα στους τρέχοντες λογαριασμούς της οντότητας αυτής είναι τα μεγαλύτερα σε ολοκληρό κόσμο και σίγουρα θα μπορούσαμε να βοηθηθούμε πάρα πολύ για να αντιμετωπίσουμε τη ζήτηση κλπ. Όμως, το να υπάρχει συντονισμός δεν σημαίνει ότι πρέπει και όλοι να είμαστε ίδιοι. Οι συστάσεις ζητούν από τις χώρες μέλη να δράσουν και συλλογικά αλλά και ατομικά για να ανταποκριθούν στις διάφορες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Κυρίως οι χώρες μέλη εκείνες που έχουν τρέχοντες λογαριασμούς που απαιτούν μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Όπως επίσης όμως και άλλες χώρες που έχουν πλεονάσματα θα έπρεπε να φροντίσουν για περισσότερες επενδύσεις. Και όλα αυτά για να αποφύγουμε την ε, τελμάτωση και να προχωρήσουμε σε μεταρρυθμίσεις. Οι χώρες που έχουν υψηλά επίπεδα δημοσίου χρέους επίσης θα έπρεπε να το μειώσουν και οι χώρες που έχουν δημοσιονομικό περιθώριο θα έπρεπε να φροντίσουν για περισσότερες υψηλής ποιότητας επενδύσεις. Επίσης, ζητάμε από τις χώρες μέλη να στηρίξουν μια δίκαια μετάβαση, χωρίς να ξεχάσουν κανέναν, για μια ανταγωνιστική πράσινη και ψηφιακή οικονομία, τόσο με επενδύσεις υλικές όσο και με υλικές. Η πράσινη ε, μετάβαση είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει πραγματικότητα. Ξέρουμε όμως πως για πολλούς εργαζόμενους είναι και μια μεγάλη δυσκολία. Πρέπει λοιπόν να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στα πλαίσια αυτού του μηχανισμού μετάβασης. Και αυτό να το πετύχουμε ε, συγχρονίζοντας ε, καλά με το πνεύμα αυτό και τις επενδύσεις για την Πράσινη Συμφωνία. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε επίση το θέμα της εταιρική φορολογίας, κάτι το οποίο παραμένει προτεραιότητα για μα. Τέλος, επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια και για την έκθεση όσον αφορά τον μηχανισμό επαγρύπνησης ε, με τον οποίο ξεκινάει ο ετήσιος κύκλος της διαδικασίας για, την για τη διαδικασία μάλλον μακροοικονομικών ανισορροπιών. Η γίνεται σε βάθος ανάλυση. Τα καλά νέα είναι ότι μόνο οι ίδιες 13 χώρες μέλη που πέρασαν την ανάλυση αυτή σε βάθος πέρυσι πρέπει να αναλυθούν εκ νέου φέτος. Επίσης η έκθεσή μας αναφέρει και διάφορα μηνύματα που έχουν να κάνουν με εξελίξεις που δεν προχώρησαν. Πρέπει να υπάρχει διόρθωση διάφορων ανισορροπιών, κυρίως εκείνων που έχουν να κάνουν με ε, μεγάλο χρέος και πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες. Επίσης, να συνεχιστούν και προσπάθειες ε, διαρθρωτικών ε, μεταρρυθμίσεων. Οι προοπτικές δεν είναι τόσο καλές, οπότε δεν ευνοούν τη συνέχεια. Εκ παραλίλου αναδύονται και νέοι κίνδυνοι, κυρίως εξαιτίας των ε, τιμών της κατοικίας που συνεχίζουν να αυξάνουν παντού, όπως επίσης και το μοναδιαίο εργασιακό κόστος, το οποίο επίσης ενισχύεται κυρίως στις χώρες κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης αλλά και στις βαλτικές χώρες. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα περάσει στο επόμενο βήμα της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών παρουσιάζοντας τις εκθέσεις σε βάθος και τις εκθέσεις αναχώρα στα τέλη Φεβρουαρίου. Εποφελούμε λοιπόν από αυτή την ευκαιρία για να επιβεβαιώσω ότι είμαστε στη διάθεσή σας για ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά τις αναχώρα συστάσεις πριν αυτές ε, δημοσιοποιηθούν ε, κάτι το οποίο θα γίνει στα τέλη Φεβρουαρίου. Είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε ερωτήσεις και δίνω το λόγο στην Πρόεδρο. Ναι, ναι, βέβαια μπορούμε να αλλάξουμε και ρόλους, γιατί όχι. Θα δώσω το λόγο τώρα στον Νίκολα Σμίτ, λοιπόν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, θα ξεκινήσω στα γαλλικά και μετά θα συνεχίσω με την αγγλική. Ε, με μεγάλη χαρά βρίσκομαι ανάμεσά σας πάλι. Η οικονομική και κοινωνικονομική διακυβέρνηση έχει σαν βασικό στόχο να ενισχύσει την κοινωνική οικονομία της αγοράς μια αγορά η οποία θα πρέπει να υπηρετεί τους πολίτες όπως το εξήγησε και η Ursula von der Για να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει να βασιστούμε ε, στα κοινωνικά δικαιώματα. Ξεκίνησε μια συζήτηση δηλαδή από τις 14 Ιανουαρίου για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να ενισχύσουμε την κοινωνική Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε επίσης και τα πρώτα στοιχεία ενός πλαισίου για ένα ελάχιστο μισθό για το σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκινώντας με το έδαφος θα έλεγα για μία πρώτη διαβούλευση. Η ετήσια στρατηγική για μία αηφόρο ανάπτυξη έχει σαν στόχο την προώθηση μιας οικονομίας που συνδυάζει την αγορά, την, οικονομική σταθερότητα, την κοινωνική προστασία και την καταπολέμηση των συνεπειών του, ε, του κλίματος. Τώρα, η ενίσχυση του κοινωνικού πολέ, ε, πυλώνα θα βελτιώσει την ανθεκτικότητα της οικονομίας μας και θα προωθήσει τη σύγκληση και την καινοτομία. Αυτό είναι αλήθεια σε έναν τομέα τόσο προχωρημένο και ολοκληρωμένο όπως η νομισματική ένωση. Η οικονομική σύγκληση και η κοινωνική σύγκληση θα πρέπει να συμβαδίζουν. Και γι' αυτό οι προτάσεις, οι συστάσεις μάλλον αναχώρα, κάνουν προτάσεις σε σχέση με τους πυλώνες όπως η ενίσχυση των επενδύσεων στην παιδεία, στην κατάρτιση, στις πολιτικές της αγοράς εργασίας, προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και διασφάλιση της ισότητας φύλων σε όλα τα επίπεδα. Καταρχάς, δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης και αποτροπή διάσπασης της αγοράς εργασίας, πόλη διάσπασης της αγοράς εργασίας, ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου και των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Φέτος η πρόταση για την κοινή έκθεση δείχνει ότι η Ευρώπη έχει κάνει πρόοδο και στον τομέα των κοινωνικών δικαιωμάτων. Η απασχόληση αυξάνεται. Ε, αυτή τη στιγμή ε, απασχολούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση άνω των 200 ε, εκατομμυρίων εργαζομένων, κάτι το οποίο αποτελεί το υψηλότερο, αν θέλετε, ποσό εργαζομένων που έχει σημειωθεί ποτέ. Όμως, τα, οι ανισότητες σε επίπεδο εισοδημάτων παραμένουν σε υψηλό επίπεδο και σε διαφορετικούς τομείς όπως η βελτίωση ε, των ικανοτήτων, οι ε, μισθολογικές και φορολογικές διευκολύνσεις και κίνητρα, διασφάλιση ε, σε προσβάσιμες κοινωνικές υπηρεσίες και στον τομέα της κατοικίας και κυρίως προώθηση, επίσης μάλλον προώθηση ισότητας ευκαιριών. Οι διαφορές στις ε, αμοιβέ ανδρών γυναικών είναι στο ίδιο σχεδόν επίπεδο από το 2013. Έγιναν κάποια βήματα προόδου το 2018, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει επίσης το ύψος των μισθών να συνδυάζεται με τη βελτίωση της αποδοτικότητας. Ε, η εσωτερικοί θύλακοι φτώχειας παραμένουν ιδιαίτερα σε νοικοκυριά τα οποία εργάζονται με προσωρινές ή άτυπες σχέσεις εργασίας. Στις 4 Μαρτίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταθέσει μια νέα ατζέντα για την απόκτηση ικανοτήτων επαγγελματικών που θα βοηθήσει τους εργαζομένους να ακολουθήσουν τις αλλαγές της αγοράς εργασίας και τις αλλαγές στο περιβάλλον και στην μετάβαση στη νέα κατάσταση. Συνεχής βελτίωση των ικανοτήτων και απόκτηση νέων δυνατοτήτων. Έτσι θα βρεθούν νέες θέσεις εργασίας, έτσι θα αμφισβητηθούν στρεβλές πρακτικές και θα εγκαταλειφθούν πρακτικές οι οποίες δεν είναι προσαρμοσμένες στις νέες ευκαιρίες. Βασικός στόχος είναι να δώσουμε κοινωνική προστασία σε όλους τους εργαζομένους ανεξαρτήτως του επίπεδου απασχόλησής τους. Τα κοινωνικά συστήματα πρέπει να εξυγχρονιστούν. Υπάρχουν όμως κατηγορίες επαγγελματικές που έχουν θέματα όπως οι αυτοαπασχολούμενοι. Επίσης ε, υπάρχουν θέματα με τα συστήματα κοινωνικής προστασίας είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητηθεί ακόμα περισσότερο. Πρέπει να προωθηθεί επίσης η αηφορία και η βιωσιμότητα της μακροπρόθεσμης φροντίδας και να αντιμετωπιστεί και το θέμα της ανεπίσημης φροντίδας. Τώρα για τον τελευταίο πυλώνα έχει υπάρξει πρόοδο στα πλαίσια της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του εθνικού επίπεδου και των τοπικών αρχών και της κοινωνίας των πολιτών. Η εφαρμογή των πυλώνων αυτή είναι θα έλεγα μεικτή αρμοδιότητα της Ένωσης και των υπολείπων όλων και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μεταφέρει τις απόψεις τους, τις οποίες υπολογίζουμε γιατί είναι εκπρόσωπος των λαών της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ακούσουμε τον πρώτο γύρο ερωτήσεων. Όπως κάνουμε συνήθως, θα ξεκινήσουμε ε, από τους εισηγητές της ΕΚΟΝ και της ΕΜΠΛ για τις ε, εκθέσεις ε, αυτές του εξαμήνου και κατόπιν θα ακούσουμε τις απαντήσεις των Επιτρόπων Δύο λεπτά ο καθένας θα έχει για να απαντήσει. Δίνω το λόγο στην κυρία Γολαλίκ ε, από την ΕΚΟΝ. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω γαλλικά. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί επίτροποι, αγαπητοί συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε να ξαναδούμε το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Εξάλλου αλλάζω τίτλος του της έκθεσης που μιλάει για ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην έκθεση που έχω αναλάβει εγώ και που θα αρχίσουμε να διαπραγματευόμαστε σύντομα, υπάρχει αυτή η νέα ε, προσέγγιση μέσω αλλαγής δικτών και μέσω της ε, ένταξης και των ε, στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Ξέρουμε βέβαια ότι το βασικό είναι οι δημόσιες δαπάνες προκειμένου να πετύχει η οικολογική μετάβαση γιατί ο ιδιωτικό κλάδος δεν θα μπορέσει να αντικαταστήσει το δημόσιο και στο κάτω-κάτω δεν είναι καν αυτός ο ρόλος του. Τελευταία διαπιστώνουμε στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Πολωνία, στην Ισπανία σε διάφορους κλάδους ότι δεν υπάρχουν αρκετές επενδύσεις ούτε για τις ανώσιμε πηγές ενέργειας ούτε για τις υποδομέ. Όλοι λοιπόν έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο ε, χαμηλών επενδύσεων. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι απλή. Κατά τη διάρκεια της δημοσιονομικής κρίσης ξεπεράσαμε ένα ταμπού στην Ευρώπη που ήταν εκείνο της χρησιμοποίησης της νομισματικής πολιτικής. Τώρα η οικολογική κρίση θα μας βοηθήσει επίσης να γίνουμε ρεαλιστές και να ξεπεράσουμε ένα άλλο ταμπού που είναι εκείνο των δημοσίων δαπανών. Δηλαδή θα ήθελα να ξέρω τη γνώμη σας ε, τόσο όσον αφορά το χρυσό κανόνα δηλαδή οι δαπάνες που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον να μην υπολογίζονται ε, αρνητικά στις δημόσιες δαπάνες και έπειτα ε, για την αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας ε, και Ανάπτυξης των δύο οδηγών και των έξι οδηγιών. Ακούσαμε ότι δεν μπορεί να υπάρχει οικονομική πολιτική αποτελεσματική χωρίς αναθεώρηση των δύο αυτών πακέτων. Οι φιλοδοξίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μεγάλε για να απαλλαγεί Ευρώπη από τον άνθρακα. Εμεί χαιρετίζουμε αυτή τη φιλοδοξία, η οποία όμω πιστεύω ότι δεν θα πετύχει αν δεν ξεπεράσουμε τους δημοσιονομικούς περιορισμούς. Γι' αυτό θα ήθελα τη γνώμη σα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Κλάρα Ντόμπρεφ, εκ μέρου τη Επιτροπή Απασχόληση. Ευχαριστώ πολύ. Όπω είπατε, κύριε Ντομπρόφσκι, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αντιμετωπίσει και οικονομική ανάπτυξη τα τελευταία δέκα χρόνια. Έχουμε καλά στοιχεία. Αν δούμε τις επενδύσεις, ΑΕΠ, απασχόληση και άλλους μακροοικονομικούς δείκτες, ε, τα αποτελέσματα είναι θετικά σε Υψη ρεκόρ μερικές φορές. Αυτή όμως είναι η μία πλευρά του νομίσματος, γιατί υπάρχει και η άλλη, η οποία δεν είναι τόσο λαμπρή. Παρά το μέσο όρο ανάπτυξη, οι ανισότητες στι κοινωνίε μας στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει φτώχεια, φτώχεια των παιδιών για παράδειγμα, κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό και αυξάνει και βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Και η κατάσταση δεν φαίνεται να βελτιώνεται παρά τα ωραία οικονομικά στοιχεία, παρά ε, τα στοιχεία για την ετήσια ανάπτυξη, παρόλα αυτά στα κοινωνικά δεν τα καταφέρνουμε. Και δεύτερον, συζητάμε πολύ για τις προκλήσεις, για την κλιματική αλλαγή και έχουμε αναλάβει κάποια βήματα που ελπίζω να φτάσουν. Αλλά δεν πρόκειται να φέρουμε σε πέρας αυτά που θέλουμε αν δεν φέρουμε με το μέρος μας ε, τους εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες. Υπάρχει δηλαδή και η κοινωνική πτυχή της Πράσινης Συμφωνίας που δεν θα πρέπει να τη βλέπουμε σαν κάτι απ' έξω. Όχι σαν κάτι που πρέπει να κάνουμε έτσι για να είμαστε καλά. Όχι, πρόκειται για την καρδιά της Πράσινης Συμφωνίας. Χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη, χωρίς ισχυρές κοινωνικές πτυχές δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε τις υποσχέσεις που δώσαμε για την Πράσινη Συμφωνία και δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε στους εαυτούς μας να αποτύχουμε. Συνεπώς, χρειαζόμαστε ένα νέο μοντέλο, ένα νέο πρότυπο. Κύριε Ντομπρόφσκι, είπατε ότι πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη και βιωσιμότητα. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι η βιωσιμότητα σημαίνει οικονομική βιωσιμότητα, κοινωνική βιωσιμότητα και οικολογική βιωσιμότητα. Τρία σε ένα. Σε ένα όμως. Δεν μπορούμε να τα χωρίσουμε το ένα από το άλλο. Μερικές φορές μιλάτε για τη δικαιοσύνη σαν να είναι κάτι επιπλέον που πρέπει να φροντίσουμε δίπλα στην ε, ε, βιώσιμη οικονομική μας πολιτική ή το περιβάλλον. Όχι. Είναι ένα με τα υπόλοιπα. Πώς λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διασφαλίσει η δικαιοσύνη, όπως είπατε κι εσείς, να είναι μέρος του νέου μοντέλου, εξίσου σημαντική με τα υπόλοιπα όσον αφορά τις επενδύσεις και να έχουμε κατάλληλες επενδύσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στον κύριο Ντομπρόφσκης, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας αυτές. Σας ξεκινήσουμε λοιπόν από την πρώτη ερώτηση για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Πράγματι, Εάν κάνετε τη σύγκριση με την προηγούμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα διαπιστώσετε ότι αλλάξαμε το αφήγημα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου σε σημαντικό βαθμό. Γι' αυτό αλλάξαμε και τον τίτλο του εγγράφου. Η ετήσια επισκόπηση ανάπτυξη. γίνεται ετήσια στρατηγική βιώσιμη ανάπτυξη για να αντικατοπτρίσουμε το νέο αυτό αφήγημα, το νέο τρόπο να εξετάζουμε οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά, κλιματικά ε, στοιχεία με ολοκληρωμένο και ολιστικό τρόπο. Αυτό λοιπόν αποτελεί την βάση για την προσέγγιση μας όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Όσον αφορά τις ερωτήσεις σχετικά με την αναθεώρηση ε, το, της δέσμης 2 μέτρων και δέσμης 6 ε, μέτρων αντίστοιχα. Αυτή τη στιγμή ε, ετοιμα, ετοιμαζόμαστε για την αναθεώρηση αυτή. Εξετάζουμε τους δημοσιονομικούς μας κανόνες, ενώ παράλληλα σκοπεύουμε να ξεκινήσουμε δημόσια διαβούλευση με ανοιχτό τρόπο, χωρίς να προδικάζουμε το αποτέλεσμα, για να εξετάσουμε προς ποια κατεύθυνση πρέπει να πάμε με τους δημοσιονομικούς κανόνες. Μετά τη δημόσια αυτή διαβούλευση θα επανέλθουμε και θα σας προτείνουμε τα επόμενα βήματα. Όσον αφορά την ουσία, μπορεί να είναι ακόμη πολύ νωρίς να εξάγουμε συμπεράσματα, αλλά Νομίζω ότι και η συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου σχετικά με τους ε, κανόνες, ε, τα σημεία αναφοράς ε, και τον περιορισμένο χρυσό κανόνα, νομίζω ότι αυτά θα αποτελέσουν αφετηρία για συζήτηση. Συζητώντας τη βιωσιμότητα και τις επενδύσεις, θα ήθελα να ε, τονίσω τη σημασία του ε, επενδυτικού σχεδίου της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Ο στόχος μας είναι να συγκεντρώσουμε ε, τουλάχιστον ένα τρισεκατομμύριο βιώσιμων επενδύσεων την επόμενη δεκαετία. Κατόπιν ήθελα να πω ότι οι κοινωνικές στοιχές αποτελούν τμήμα του νέου αφηγήματός μας. Εξετάζουμε όλα αυτά τα θέματα συνολικά. Αυτό ακριβώς ε, τονίζει συνεχώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι χρειάζεται να έχουμε μια πράσινη μετάβαση, να προσαρμοστούμε ε, στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, καθώς και στη γύρανση του πληθυσμού, με τρόπο κοινωνικά αποδεκτό που να διατηρεί ε, το ε, πρότυπό μας, ε, το μοντέλο της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. Θα ήθελα επίσης να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι μόλις εκδώσαμε ανακοίνωση για μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Τζεντιλόνη. Να απαντήσω στην ερώτηση της κυρίας Λαλούκ. Οι λέξεις που χρησιμοποίησε η πρόεδρος Φοντερ Λάιεν είναι ακριβώς ε, αυτές όταν είπε ότι η Πράσινη Συμφωνία είναι η νέα μας στρατηγική ανάπτυξης. Και πιστεύω ότι υπάρχει ένα μήνυμα μέσα σε αυτά τα λόγια. Πρέπει να δουλέψουμε ε, πάνω σε αυτό, όπως το είπε μόλις και ο Βάλτης. Θα επανακινήσουμε και τη διαδικασία αναθεώρησης των πακέτων των έξι οδηγιών και των δύο οδηγιών και στα πλαίσια αυτά δεν έχουμε αμέσως κάποια λύση, χρειάζονται μήνες συζήτηση και σίγουρα θα συμμετέχει πλήρως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι στόχος μας είναι οι δημόσιες επενδύσεις και οι ιδιωτικές επενδύσεις να καταστούν πιο εύκολες. Αυτό είναι ο στόχος. Γιατί σαφώ και υπάρχει μια κατάσταση όπου δεν έχουμε αρκετές επενδύσεις. Για τον, την κυρία Ντόμπρεβ. Συμφωνώ μαζί σας για το ότι όταν συζητάμε για βιωσιμότητα χρησιμοποιούμε μια γενική ιδέα και αντίληψη για τη βιωσιμότητα που έχει να κάνει με το περιβάλλον, αλλά έχει να κάνει και με τα κοινωνικά ε, δικαιώματα. Και η εμπειρία μας από την ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια μας ε, οδηγεί να θέλουμε να μην υπάρχουν κοινωνικές συνέπειες. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να συμπεριλάβουμε δηλαδή στο ευρωπαϊκό εξάμεινο και τις κοινωνικές πτυχές και τις περιβαλλοντικές πτυχές χωρίς όμως βέβαια να περιορίζουμε τον μακροοικονομικό ορίζοντα. Νομίζω ότι μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ, ο κύριος Σμιτ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να, να προσθέσω κάτι κι εγώ σε αυτά που είπε ο κύριος Τζεντιλόνε. Είναι σαφές ότι η κοινωνική διάσταση είναι εξίσου σημαντική σε αυτήν την μετάβαση, σε αυτές τις μεταβάσεις, γιατί έχουμε την πράσινη, αλλά έχουμε και την ψηφιακή μετάβαση. Συνήπως, έχουμε μια ανακοίνωση που λέγεται «Η ισχυρή Ευρώπη για δίκαια μετάβαση». Και το εργαλείο που έχουμε είναι βέβαια η υλοποίηση του, κοινού, του κοινωνικού πυλώνα. Έπειτα είναι η επένδυση στον άνθρωπο. Δηλαδή όταν μιλάμε για επενδύσεις, να μιλάμε και για επενδύσεις πάνω στον άνθρωπο, τις δεξιότητες του ανθρώπου, για παράδειγμα. Έτσι θα πετύχουμε τη δίκαια μετάβαση για όλους, χωρίς να ξεχάσουμε κανέναν. Έπειτα, το να δημιουργήσουμε, να επενδύσουμε δηλαδή και να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης ποιότητα, αγορά εργασίας. Και αυτά είναι στοιχεία κλειδιά, επειδή συζητούμε για τους μισθούς στην Ευρώπη, για ένα πλαίσιο ελάχιστου μισθού ή για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων, την καταπολέμηση της φτώχειας, το είπατε κι εσείς. Η φτώχεια των παιδιών αποτελεί κεντρικό στοιχείο σε αυτά που συζητάμε και ε, σχεδιάζουμε επίσης και μία εγγύηση για τα παιδιά. Περνάμε στο δεύτερο γύρο, έχουμε τέσσερις ομιλητές, ο κάθε ένας θα έχει 1,5 λεπτό. Ράτκε. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπη, ε, θα ήθελα καταρχά να ευχαριστήσω τους επιτρόπους που βρίσκονται εδώ για να μας απαντήσουν ε, στις ερωτήσεις μας. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Βάλτη που ε, στην εισήγησή του αναφέρθηκε στην κοινωνική δικαιοσύνη και είπε ότι βρίσκεται στον πυρήνα της πολιτικής δουλειά τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Πολύ συγκεκριμένη ερώτηση λοιπόν θα ήθελα να θέσω όσον αφορά το Ταμείο Δικαίη μετάβαση αναφέρεται, συζητιέται το πώς διαμορφώνεται. Θα ήθελα να τονίσω ότι βρίσκω θεμελιώδους σημασία σε ένα τέτοιο ταμείο. Ε, αλλά ε, θα, δεν θα μπορούσα ποτέ να δεχτώ να γίνει αυτό εις βάρος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Η πράσινη μετάβαση της οικονομίας μας είναι απολύτως απαραίτητη, αλλά δεν επιτρέπεται αυτό να γίνει η βάρος άλλων ε, μειονεκτικών ομάδων ε, στα κράτη-μέλη μας. Και γι' αυτό θα ήθελα να ε, σχολιάσετε το θέμα αυτό. Και μία ερώτηση προς τον κύριο Σμιτ. Ε, που θα ασχοληθεί κατά τη διάρκεια του έτους με το θέμα του ελάχιστου μισθού. Η διαδικασία ήδη έχει ξεκινήσει. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι άσχετα από το πώς θα καταλήξει η διαδικασία αυτή, όσον αφορά τις ε, συλλογικές συμβάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλάμε για την ανάπτυξη, μιλάμε για ε, τα πόσα έχει προσφέρει αυτά στο πορτοφόλι του, ε, ε του εργαζόμενου. Ε, τα τελευταία 30 χρόνια στη Γερμανία, για παράδειγμα, στη χημική βιομηχανία είχαν αύξηση οι εργαζόμενοι 30%. Ε, θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω να σχολιάσετε το θέμα αυτό. Ο Μάρκους Φέρμπερ από την Επιτροπή ΕΚΟΝ από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω και εγώ γερμανικά, ε, αν μου το επιτρέπετε. Θα προσπαθήσω στο σύντομο χρονικό διάστημα που δίνεται να παρουσιάσω τις παρατηρήσεις μου και να επικεντρωθώ στο θέμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι θέλει να κάνει πιο λιτό το εξάμεινο, να έχει λιγότερες συστάσεις αναχώρα ε, και να έχει σαφείς στόχους ε, επενδύσεις, διαφορετικές μεταρρυθμίσεις και διασφάλιση μιας ε, υπεύθυνης δημοσιονομικής πολιτικής. Ε, στην ε, στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης 2020, το τρίγωνο αυτών των στόχων έχει γίνει τετράγωνο διότι έχουμε και μια πολύ θολή διάσταση περιβάλλον, παραγωγικότητα κλπ. Έχουμε λοιπόν τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, οι οποίοι θα πρέπει να ενσωματωθούν στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Εγώ λοιπόν αναρωτιέμαι, εσείς πώς βλέπετε την ενσωμάτωση των στόχων αυτών και πώς αυτό ταιριάζει με τον πρόσφατα διατυπωμένο στόχο ενός ε, πιο στοχευμένου ευρωπαϊκού εξαμήνου, όπως ζητάει το Κοινοβούλιο σε πολλά ψηφίσματα τα τελευταία χρόνια. Εμένα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα ο στόχος 8 των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Πώς θα ενσωματωθεί αυτό στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μαρία Πιέρ από την Επιτροπή ε, ΕΜΠΛ. Θέλω να σας ευχαριστήσω, Επίτροπη, για την παρουσία σας σήμερα εδώ και για τις απαντήσεις σας. Η παρουσία σας δείχνει ότι η δημοκρατική ευθύνη και η οικονομική και κοινωνική διακυβέρνηση συμβαδίζουν. Πράγματι καλά κάνετε και υιοθετήσατε το, το πράσινο σύμφωνο ουσιαστικά στις οικονομικές σας και κοινωνικές προτάσεις. Οι δηλώσεις αυτές όμως δεν πρέπει να παραμείνουν γράμμα νεκρό. Μιλήσατε για πρωτοβουλίες όπως ο ελάχιστος μισθός και οι ψηφιακές αρμοδιότητες. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις προτάσεις σας στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, ιδιαίτερα σχετικά με την απασχόληση, που πολλές φορές τα ξεχνάμε γιατί επικρατεί ο προϋπολογισμός. Δύο ερωτήσεις. Στη στρατηγική σας δεν αναφέρεστε στην κινητικότητα των εργαζομένων, ενώ στην προηγούμενη περίοδο είχαν υπάρξει αρκετές πρωτοβουλίες. Τι μέτρα λοιπόν θα πάρετε για να διασφαλίσετε την κινητικότητα των εργαζομένων που θα πρέπει να είναι δίκαιοι και δεύτερη ερώτηση αφορά το κοινωνικό ταμείο, το Ταμείο ε, ε, Δίκαιης Μετάβασης και το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση. Στόχος είναι να πετύχουμε αυτή τη μετάβαση στον τομέα τον ψηφιακό και στον τομέα τον κλιματολογικό πώς θα διασφαλίσετε τη συνοχή αυτών των ε, ταμείων. Ο κύριος Ερόγλου από την Εκόνα, Ρινιού. Κυρία Πρόεδρε, κύριοι Επίτροποι, σας ευχαριστούμε για τη δυνατότητα που μας δίνετε σήμερα να σας θέσουμε ερωτήσεις. Θα ήθελα να παραθέσω λόγια του ε, Ομοσπονδιακού Υπουργού Οικονομικών μας, ε, σας τα διαβάζω, τα έχω κατεβάσει από το ίντερνετ ε, και αναφέρεται στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Λέει ότι στα περιθώρια αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, σε κάθε ε, αρχή έτους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει μία ε, έκθεση ανάπτυξης. Αναφέρονται οι συστάσεις που δίδονται στα κράτη-μέλη. Ο ομοσπονδιακό Υπουργό Οικονομικών ε, δεν ανήκει στο δικό μου πολιτικό στρατόπεδο, αλλά συμμερίζομαι απόλυτα τι παρατηρήσει του, διότι πιστεύω και εγώ ότι έχει αλλάξει ο στόχος της έκθεσης αυτής. Ε, και ε, γι' αυτό θα ήθελα να θέσω την εξή ερώτηση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι σημαντικό να λαμβάνουμε αποφάσει σχετικά με τα μεταρρυθμίσει, αλλά ε, είναι εξίσου σημαντικό να ε, εφαρμόζονται από τα κράτη-μέλη. Έχω τι ίδιε ανησυχίε με τον συνάδελφο από το ΕΛΚ. Αν επιβάλλουμε άλλη μια δέσμη μέτρων, ε, ε, φοβάμαι ότι δεν θα πραγματοποιηθούν οι σημαντικέ μεταρρυθμίσει. Ερώτηση λοιπόν προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει αλλάξει το επίκεντρο, δεν μιλάμε πια για διορθωτικέ μεταρρυθμίσεις. Μας απασχολεί περισσότερο η έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης ε, στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Σας ευχαριστώ. Very Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα πάρουμε τις απαντήσεις από τους τρεις επιτρόπους. Ο κύριος Ντομπρόφσκης πρώτος. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητά μέλη. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Τώρα για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το πώς συνδέεται με το ε, ESF+, το κοινωνικό συν. πως οι προτάσεις αυτές θα ξεπεράσουν το 1,11% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ που εμείς προτείνουμε. αυτή η συζήτηση η οποία ψάχνει να δώσει απαντήσεις στα αν αυτές οι προτάσεις θα είναι εις βάρος του κοινωνικού ταμείου ή του ταμείου συνεχής πρέπει να σταματήσουν. Εμείς ζητάμε επιπλέον χρήματα. Το κοινοβούλιο είναι ακόμα πιο φιλόδοξο, θέλει και μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ αλλά οι συζητήσεις στο Συμβούλιο προς το παρόν θεωρούν ότι ήδη το 1.11 είναι πολύ υψηλό. Η συζήτηση δεν θα είναι πολύ εύκολη. Οι προτάσεις της Επιτροπής θα πρέπει όμως να είναι υπεράνω των ποσών που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας, των ποσοστών συγγνώμη, που έχουμε στη διάθεση. Τώρα για το εξάμεινο και το streamlining του εξαμήνου. Στον τομέα αυτό δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν κάποιες επιπλέον συστάσεις σε τομείς όπως ε, η φροντίδα και τα μέτρα τα οποία προβλέπονται και τα ταμεία για τους νέους. Ο στόχος μας θα είναι τα μακροοικονομικά και τα κοινωνικά, εντάσσοντας όμως την προτάσεις αυτές και την αηφορία. Θα πρέπει φυσικά πάντα να λαμβάνουμε υπόψη μας την αξιολόγηση των επιδόσεων των κρατών μελών και το πόσο εντάσσουν τους στόχους της αηφορίας. Γενικά όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους και όλα συναποτελούν το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο έτσι ώστε ε, να προχωρήσουμε σε, ε, προς την πορεία της βελτίωσης των θέσεων απασχόλησης και της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης, βασικός στόχος του κάθε εξαμήνου. Τώρα για την ετήσια στρατηγική και τις διαφορετικές αλλαγές. Ε, πράγματι παραμένει η προσοχή την οποία δίνουμε εμείς στις διαφορετικές αλλαγές. Ε, προώθηση φυσικά της ανταγωνιστικότητας. Εδώ είναι απαραίτητες οι ε, διαφορετικές αλλαγές. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Επίτροπος Τζεντιλόνι. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά τα οποία είπε ο ε, για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Η πρότασή μας είναι σαφής και τα χρήματα για το Ταμείο αυτό θα πρέπει να προέλθουν επιπλέον των ήδη υπαρχουσών δυνατοτήτων. Πάντα για το εξάμεινο πρέπει να πούμε ότι ο στόχος για να γίνουν τα πράγματα με κάπως πιο απλή τρόπο, που είναι καλός στόχος, δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι ε, δεν μπορούμε να έχουμε κάποιους άλλους στόχους. Ήδη έχουμε τον κοινωνικό τομέα, ήδη έχουμε τον πίνακα επιδόσεων, το social scoreboard. Και εμείς έχουμε μιλήσει πάρα πολύ σήμερα για την αηφορία, για το περιβάλλον, για τους στόχους συμπερίληψης, διότι εδώ αν θέλετε έχουμε να κάνουμε με μια νέα ρητορική η οποία επιβάλλεται και η οποία καθορίζει την πολιτική μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μειώσουμε το βάρος που δίνουμε στις διαφθορτικές αλλαγές και στις μακροοικονομικές ανισότητες. Θα μπορέσουμε πράγματι τώρα να απλοποιήσουμε τον μηχανισμό αυτό τον οποίο έχουμε στη διάθεσή μας. Η συζήτηση την οποία είχαμε μέχρι τώρα μεταξύ μας και με τα κράτη-μέλη και ε, που φαίνεται και στην έκθεση ε, του European Fiscal Board, το μήνυμα της απλοποίησης δεν είναι τόσο ένα μήνυμα που λέει μην προσθέτετε άλλα θέματα για συζήτηση. Είναι ένα θέμα απλοποίησης του μηχανισμού που έχει στόχο την αντιμετώπιση και τη μείωση των μακροοικονομικών ανισοτήτων ανισορροπιών περισσότερο. Ε, πρέπει λοιπόν εμείς ε, να μην παραβλέψουμε τον βασικό στόχο. Καταλαβαίνω αυτούς οι οποίοι φοβούνται μια διάχυση, μια πολυδιάσπαση. Θα ήθελα να πω ότι στον κύριο Φέρμπερ ότι το 8 σαν παράδειγμα εντάσσεται ήδη στον κοινωνικό πυλώνα Υπάρχουν και στόχοι άλλοι από την αηφορία που έχουν σχέση με το κράτος δικαίου, έχουν σχέση με τη δικαιοσύνη και δεν εντάσσονται από μόνα τους αυτόματα στο ε, εξάμεινο. Ε, θα πρέπει να τα εντάξουμε στα πλαίσια του νέου προγραμματός μας. Ο στόχος λοιπόν της απλοποίησης είναι ένας σαφέστατος στόχος, Νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή ε, κρατώντας το νου μας ε, και τον κοινωνικό τομέα και τον περιβαλλοντικό τομέα σε συνδυασμό με όλα τα προηγούμενα. Ευχαριστώ. Ο τρίτος επίτροπος, ο κύριος Σμιτ. Θα ομιλήσω γερμανικά, πρόεδρε, για το πρώτο τμήμα δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποια σύγχυση ή κάποια σύγκρουση ανάμεσα στο κοινωνικό ταμείο πλάσα και στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Νομίζω ότι και τα δύο μπορούν να συνεργαστούν. Ξέρουμε ότι δεν έχουμε την πανάκια στην διάθεσή μας, αλλά βοηθάει να μπορέσουμε να αυξήσουμε ας πούμε λίγο, τους, να κινηθούν λίγο οι αμοιβέ αλλά ο στόχος εκεί είναι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις. Και σε πολλές χώρες δεν υπάρχουν επαρκώς κοινωνικές, τέτοιες συλλογικές διαπραγματεύσεις, τουλάχιστον σε, οικονομικό, σε ικανοποιητικό επίπεδο. Θα πρέπει οι κοινωνικές αυτές διαδικασίες να αποκτήσουν μια νέα όθηση. Εκεί όπου υπήρχαν ισχυρές συλλογικές διαπραγματεύσεις, στους τομείς αυτούς η κατάσταση έχει κάπως βελτιωθεί. Αν και υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις και αναφέρουμε εδώ περισσότερο στη Γαλλία τώρα για το ODD8 δηλαδή τους στόχους της αριφορίας σε σχέση με τις θέσεις απασχόλησης. Κοιτάξτε, στόχος μας είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης καλής ποιότητας, ικανοποιητικής ποιότητας. Γιατί έχουμε ανάγκη από τέτοιες θέσεις. Γιατί έτσι θα μπορέσουμε να ενταχθούμε σε ένα νέο κύκλο ανάπτυξης, σε μια νέα στρατηγική ανάπτυξης. Και έρχομαι εδώ στα λόγια του συναδέλφου Τζεντιλόνη. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το ODD 8 εντάσσεται κάλλιστα στο, στο στόχο γενικότερα για την αηφορία. Δεν υπάρχει αντίφαση σε επίπεδο ορολογίας ανάμεσα στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις από τη μία και την βιωσιμότητα από την άλλη. Αν δεν καταφέρουμε να αλλάξουμε κάποια χαρακτηριστικά μας, τις δομές μας, τότε ε, θα έχουμε φτάσει στα όρια ε, θα έλεγα των δυνατοτήτων μας. Τώρα θέλουμε να εμφαρίνουμε, λέει γαλλικά την κινητικότητα των εργαζομένων η οποία όμως θα πρέπει να είναι συμβατή με τους κοινωνικούς κανόνες και με τον κοινωνικό πυλώνα. Το κοινωνικό dumping θα πρέπει να καταπολεμηθεί με κάθε μέσο. Υιοθετήσαμε εδώ και δύο χρόνια μια οδηγία για τις αποσπάσεις των εργαζομένων. Θα τεθεί σε ισχύ στο τέλος του χρόνου και θα πρέπει η οδηγία αυτή και θα το φροντίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όχι μόνο να μεταφερθεί στις εθνικές νομοθετικές ρυθμίσεις αλλά και να αφαρμοστεί και θα φροντίσει και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Απασχόλησης. Τώρα για το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση. Ήδη από τώρα εμείς εφαρμόζουμε συγκεκριμένες ρήτρε αν θέλετε, για την ενίσχυση της ωφέλειας του Ταμείου αυτό. Ευχαριστούμε. Η πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης θα πάρει τώρα το λόγο, κύριε Λαγκελίμπελ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Τινάλη. Είμαστε στο τρίτο γύρο. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία όπως και πριν. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Σμιτ για τις απαντήσεις του. Φίλιπ ε, Λαμπέρτας, Παράκαμπ Ντονάτο και Λέση. 1,5 λεπτό η κάθε παρακαλώ και μετά θα ακούσουμε τους επιτρόπους για την απάντησή τους. Παρακαλώ, Φιλίπ Λαμπέρτ. Ευχαριστώ και καλησπέρα αγαπητή Επιτροπή. Δεν είναι μυστικό ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ που βλέπουμε νέο προσανατολισμό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και την Πράσινη Συμφωνία θεωρείται ότι είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες για τα επόμενα πέντε χρόνια. Συγχαρητήρια γι' αυτό. Θέλουμε να σας στηρίξουμε. Όμως έχουμε ένα διπλό πρόβλημα. Γιατί από τη μία γνωρίζουμε ότι δεν θα βρούμε εύκολα χρήματα για να χρηματοδοτήσουμε τις επενδύσεις που χρειάζονται. Και από την άλλη γνωρίζουμε επίσης ότι ενώ υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι στις συνθήκες, άλλοι δεν υπάρχουν. Άρα είναι και θέμα νομικής υπόστασης. Τώρα για τη διαδικασία ε, μακροπρόθεσμων ανισορροπιών. Μπορεί να αποτελεί ένα εργαλείο για να βοηθήσει στην μόχλευση και να προσανατολίσει σωστά τις πολιτικές μας. Αν δούμε το στόχο της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών, αυτό που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε είναι τις ε, αστάθειες, τις ευπάθειες των χωρών μελών μακροοικονομικά. Αν βασίζεται κανείς υπερβολικά στις εξαγωγές και σε πλεονάσματα τρεχουσών ε, συναλλαγών μπορεί να αποτελέσει μια αυπάθεια. Εξού και χαίρομαι για τη διαδικασία που λέει ότι ε, θα αναλύσουμε ακόμα περισσότερο ε, τι γίνεται με τα πλονάσματα. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο που θα μπορούσαμε να προσθέσουμε στη διαδικασία. Αν υπάρχουν υπερβολικά μεγάλες ανισορροπίες, αυτό είναι εμπόδιο για την οικονομική μεγένθηση, είναι πρόβλημα όσο περισσότερες ανισότητες έχουμε, τόσο πιο δύσκολα προχωρά η οικονομία. Που σημαίνει ότι πρόκειται για μία μακροοικονομική ευπάθεια. Αν κανείς επίσης βασίστη υπερβολικά σε ορυκτά καύσιμα και αυτό είναι λόγος ευπάθειας. Οπότε ίσως θα μπορούσατε προς αυτή την κατεύθυνση να αναθεωρήσετε τη διαδικασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ που μιλήσατε για ε, την στέγαση και τις τιμές των σπιτιών, λέει η κυρία Φαν Σπάρεντάκα, και είναι αλήθεια ότι πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να βρουν σπίτι. Έχουν αυξηθεί πράγματι τιμές σε πολλές χώρες και αυτό πρέπει να το παρακολουθήσουμε. Όμως η βασική ανησυχία της Επιτροπής είναι κυρίως η στέγαση σαν περιουσιακό στοιχείο και όχι τόσο η πρόσβαση στην στέγαση. Οπότε, κύριε Επίτροπε Ντομπρόφσκι, συμφωνείτε ότι θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί και το θέμα έλλειψης στέγασης σε ικανοποιητικέ τιμές που οδηγεί σε αποκλεισμούς και σε άστεγους. Έπειτα, Επιτροπή, μήπως θα έπρεπε εκτός από το να αναλύσει αυτές τις τάσεις, να φροντίσει να τις αντιστρέψει. Η Επιτροπή σκοπεύει να εκδώσει ειδικέ συστάσεις αναχώρα προς αυτή την κατεύθυνση και να συμπεριλάβει έναν ή περισσότερους δείχτες για το θέμα ακριβώς αυτό των τιμών της κατοικία, το πόσο κοστίζουν για παράδειγμα και πόσο αυτό πλήττει τους ανθρώπους που κινδυνεύουν να πέσουν στη φτώχεια. Τέλος, σε μεγάλες ε, ευρωπαϊκές πόλεις έχουμε ε, Airbnb και διάφορες άλλες πλατφόρμες που επίσης οδηγούν σε στεγαστική κρίση. Ε, δυστυχώς ελάχιστα μπορεί να κάνει και κάνει προς το παρόν η Επιτροπή και αποφάσεις του δικαστηρίου. Αυτό θα το θέσετε με την Επιτροπή Βαστάγκερ ώστε οι ψηφιακέ δυνατότητες να λάβουν υπόψη ότι χρειάζεται κάποια ρύθμιση και σε αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία, η κυρία Ντονάτο έχει τώρα το λόγο. Θα ήθελα να κάνω την ερώτηση και στον Τζεντιλόνι και στον Τομπρόσκης. Επανέρχομαι στο θέμα πανεξέτασης του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης έτσι ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τις συγκεκριμένες δυνατότητες, θα έλεγα, πρόκλησης του ενδιαφέροντος των επενδύσεων και έτσι να δώσουμε περισσότερες εγγυήσεις για την ανάπτυξη. Θα πρέπει να δούμε αν συμπίπτουν όμως οι λογικές μας. Είναι σαφές ε, ότι θα πρέπει να προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται με τα όρια τα οποία έχουμε σε σχέση με τα ελλείμματα του προϋπολογισμού. Ιδιαίτερα σε σχέση με τα τρέχοντα έξοδα τα οποία πολλές φορές καλύπτουν τις κοινωνικές άμεσα ανάγκες και κατά πόσον όλα αυτά συνδέονται επίσης και με το δημόσιο χρέος. Το 60% ας πούμε σε σχέση με το ΑΕΠ είναι κάτι το πάρα πολύ αυστηρό. Λίγες χώρες της Ένωσης μπορούν να σεβαστούν. Δεν υπάρχει στον κόσμο αλλού αυτό και αυτό δημιουργεί θέματα στις επενδύσεις σε χώρες οι οποίες έχουν μεγαλύτερες ανάγκες και δυνατότητες τώρα σε σχέση με αυτά τα οποία είπε ο κύριος Τζεντιλόνι. Να πω ότι αν η αποκατάσταση της ισορροπίας είναι κάτι το οποίο εγγραφεί στο χρέος των χαρών, τότε θα αναγκαστούν να μειώσουν ε, την εσωτερική ζήτηση και αυτό θα έχει προκυκλικά, θα έλεγα, αρνητικά αποτελέσματα ενώ μπορούμε να συνδυάσουμε τις προσπάθειες αυτές αν αλλάξουμε τις παραμέτρους αηφορίας ε, δημοσιονομικής. Σαν παράδειγμα ε, το Green Deal και η προσπάθεια ανέβρεσης ενός τρεις μπορεί να υπάρξει μόνο αν δημιουργήσουμε ένα κλίμα το οποίο να είναι ελκυστικό για τις ιδιωτικές επενδύσεις. ID Ευχαριστώ τους επιτρόπους για τη διαθεσιμότητά τους. Υπάρχουν θέματα πάνω στα οποία διαφωνούμε και άλλα στα οποία ζητάμε περισσότερες εξηγήσεις. Παρά την στρατηγική ετήσιας ανάπτυξης μέσω και των διαφορετικών μεταρρυθμίσεων, η κοινωνική ισότητα πάρα πολλές φορές θεωρείται από πλευρά σας δεύτερο επίπεδου θέμα. Λέτε στις προτάσεις σας ότι ε, για να προωθήσουμε την ισότητα θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τον κοινωνικό αποκλεισμό. Συνεπώς τι σημαίνει αυτό και ιδιαίτερα για κατηγορίες όπως οι αναπηρίες. Εκεί έχουν σαφώς προβλήματα και στον τομέα της απασχόλησης που πριν μερικά χρόνια δεν ξεπερνούσε το 50%. Ένας από τους δύο αναπήρους είναι άνεργος και δεν έχει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί τα ταλέντα του και τις ικανότητές του. Σύμφωνα με την έκθεση του Eurofound, το 47% ε, των αναπήρων αντιμετωπίζουν προβλήματα κατάθλιψης. Κύριε Σμιτ, τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βελτιώσει τον την κατάσταση στον τομέα της αναπηρίας ε, και πόσοι ανάπηροι εργάζονται στα ευρωπαϊκά όργανα. Τι θα κάνετε ε, σε σχέση με τις οργανώσεις των αναπήρων που ζητούν μεγαλύτερη παρουσία. Κύριε Τζεντιλόνι, στην Ιταλία εσείς μειώσατε 10 εκατομμύρια μέσα σε δύο χρόνια όταν ήσασταν υπεύθυνος για τα οικονομικά. Πώς μπορούμε να ελπίζουμε έτσι την ένταξη των αναπήρων στην οικονομία. Και κύριε Τζεντιλόνι, η απασχόληση είναι βασικό χαρακτηριστικό του κοινωνικού καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ. Ε, λέει πρόεδρος, ο κύριος Ντομπρόφσκης για να απαντήσει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ. Πρώτα απ' όλα για την Πράσινη Συμφωνία και για τη νομική ισχύ. Είχαμε ανακοίνωση, είχαμε και την πολιτική δέσμευση μέχρι το 2050 να μην έχουμε πια ε, άνθρακα αλλά ξέρετε ότι η Πράσινη Συμφωνία είναι και για το κλίμα και επειδή υπάρχει ως νόμικη υποχρέωση η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, αυτό ε, θα ενισχύσει την νομική ισχύ της Πράσινης Συμφωνίας. Έπειτα, για τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών. Είναι κάτι το οποίο ήδη χρησιμοποιούμε για τις περιπτώσεις που αναφέρατε και ακριβώς γι' αυτό η Γερμανία και οι κάτω χώρες, για παράδειγμα, είναι μέσα σε αυτή τη διαδικασία μακροοικονομικών ε, ανισορροπιών, επειδή έχουν ε, πλεονάσματα και γι' αυτό οι δύο αυτές χώρες είπαν ότι θα πακέτα ε, για δημόσιες δαπάνες ώστε να υπάρξει μια βελτίωση στις περιπτώσεις αυτές. Θα χρησιμοποιήσουν δηλαδή το δημοσιονομικό περιθώριο που έχουν για δαπάνες. Όσον αφορά τις ανισότητες, είναι ήδη μέρος του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Όπως θα θυμόσαστε και άλλες φορές έχουμε συζητήσει τις προτεραιότητές μας και έχουμε τονίσει την ανάπτυξη, χωρίς να ξεχνάμε κανέναν, την καταπολέμηση των ανισοτήτων και είπαμε ότι οι χώρες που έχουν μεγάλες διαφορές στα εισοδήματα θα συμπεριλάβουμε το θέμα των ανισοτήτων και στις συστάσεις μας και θα το κάνουμε αυτό και φέτος. Για το θέμα τώρα της πρόσβασης στη στέγαση. Πράγματι, το κοιτάμε και αυτό στις μακροοικονομικές ανισορροπίες, γιατί τότε, όντως μην ξεχάσετε ότι ξεκινήσαμε την κρίση ακριβώς από την κρίση των ανυπόθηκων δανείων. Οπότε φυσικά και μακροπροληπτικά μας απασχολεί. Ε, το κοιτάμε όμως και από την κοινωνική πτυχή. Για παράδειγμα, στο τελευταίο ευρωπαϊκό εξάμεινο όταν εντοπίσαμε τις επενδυτικές προτεραιότητες των χωρών μελών, συμπεριλάβαμε και την πρόσβαση σε στέγαση σε αποδεκτές τιμές. Και αυτό μάλιστα και στα πλαίσια του νέου πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Και η Επιτροπή θα συνεχίσει να δουλεύει προς αυτή την κατεύθυνση και στην αναθεώρηση των δημοσιονομικών κανόνων. Είπαμε ότι θα αναθεωρήσουμε τα πακέτα των 2 και των 6 οδηγιών. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Τζεντιλόνι τώρα. Παρακαλώ, κύριε Τζεντιλόνι. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Οι ευπάθειες, όπως είπε και ο κύριος Λαμπέρ, όντως είναι ένα σημαντικό στοιχείο στην ανάλυση μας των μακροοικονομικών ανισορροπιών. Και ασφαλώς, πέρα από την ισχύ των νομικών εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή μας, και όπως είπε και ο Βάλτης μόλις τώρα, ε, είναι κάτι που θα αντιμετωπιστεί μερικώς τουλάχιστον σε σχέση με την Πράσινη Συμφωνία στις συστάσεις μας, οι διάφορες ευπάθειες θα συμπεριληφθούν. Όχι μόνο οι ανισότητες, αλλά και το πόσο βασίζεται κανείς σε στερεά καύσιμα, αλλά και άλλες μακροοικονομικές ανισορροπίες έχουν ήδη ληφθεί υπόψη στις συστάσεις μας. Δεύτερον, σημειώνω τι για τη στέγαση και κυρίως για την ανάγκη να συζητήσουμε το θέμα των ε, πλατφορμών, των ηλεκτρονικών ε, πλατφορμών, που είναι ένα από τα ζητήματα που πράγματι θα συζητήσουμε την Τετάρτη ή Πέμπτη, έτσι κι θα έχουμε μία πρόταση από τον Ωσά για την φορολόγηση των ψηφιακών πλατφορμών. Και να απαντήσω τελικά στην κυρία Ντονάτο. Έχω την εντύπωση ότι στην παρουσία σας αποδείξατε τη μεγάλη σημασία που έχει η αναθεώρηση των κανόνων του Συμφώνου Ανάπτυξης και Σταθερότητας δεν ισχύει το ότι δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη γραμμή. Ξεκινάμε μια διαβούλευση δημόσια, μια συζήτηση για να μπορέσουμε να καταλήξουμε μετά την διαβούλευση φυσικά. Δύο πράγματα είναι σαφή εδώ. Το πρώτο είναι ότι έχουμε ανάγκη από τα πιο προσαρμοσμένα μέσα για να διευκολύνουμε τις δημόσιες επενδύσεις και το δεύτερο είναι ότι χωρίς ένα ευνοϊκό πλαίσιο προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων με συγχρηματοδοτήσεις δεν θα μπορέσουμε μόνο με τις δημόσιες επενδύσεις να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει. Για τους αναπήρους έχω την εντύπωση ότι θα απαντήσει καλύτερα ο συνάδελφος κύριος Σμιτ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σμιτ έχει το λόγο. Νομίζω ότι ο αντιπρόεδρος τον Μπρόσκης είπε για το πόσο βλέπουμε το θέμα της κατοικίας και της ικανοποιητικής κατάλληλης κατοικίας είναι κάτι το οποίο θα πρέπει με κάποιο τρόπο να ενταχθεί στο, στο ευρωπαϊκό εξάμεινο γιατί έχει οικονομικές πλευρές, έχει κοινωνικές πλευρές ακόμα και σε επίπεδο ανταγωνισμού υπάρχουν θέματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες μας. Τώρα για την ψηφιοποίηση να επιβεβαιώσω ότι εμείς συνεργαζόμαστε μαζί με την Αντιπρόεδρο Βέσταγκερ, ασχολούμεθα με το κοινωνικό κομμάτι της ψηφιακής ατζέντα, με τις συνθήκες εργασίας και με την κοινωνική προστασία των εργαζομένων στους τομείς αυτούς. Δεν θα αγνοήσουμε εμείς τα θέματα αυτά. Τώρα για τις αναπηρίες. Πρώτον, θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η παρούσα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει την ισότητα για όλους σε όλα τα επίπεδα. Έτσι είπε η πρόεδρος της Επιτροπής. Αυτό ισχύει λοιπόν πριν από οτιδήποτε άλλο και στους ανθρώπους με αναπηρίες. Η Επίτροπος Ντάλι θα εργαστεί για μια νέα στρατηγική για την κατάργηση των διακρίσεων εις βάρος των αναπήρων. Έχω την εντύπωση ότι μπορούμε εμείς εδώ να εντάξουμε κάποια ειδικά μέτρα για νέους αναπήρους ε, και στις ρυθμίσεις για τους νέους για να βρούνε θέση απασχόληση, για να αποκτήσουν περισσότερες ικανότητες θα πρέπει να υπάρξουν ειδικέ ρυθμίσεις για τη βοήθεια των ανθρώπων με αναπηρίες σε νεότερες ηλικίε. Ο αποκλεισμό των ανθρώπων αυτών από την αγορά εργασίας πολλές φορές συνδέεται, όχι αποκλειστικά, αλλά πάρα πολλές φορές συνδέεται ότι οι άνθρωποι αυτοί μερικές φορές δεν έχουν ικανοποιητικό επίπεδο κατάρτισης. Και αν δούμε τα μέτρα τα οποία οφείλουν να λάβουν τα κράτη-μέλη για να διευκολύνουν τη συμπερίληψή τους στην εσωτερική αγορά, ε, έχουν γίνει αρκετά. Έχουμε λοιπόν κάποια μέσα τα οποία πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα κράτη-μέλη για να ενισχύσουν και να βελτιώσουν την ικανότητα των εργοδοτών να απασχολούν περισσότερους αναπήρους. Ευχαριστώ κύριε Σμιτ. Περνάμε στον τέταρτο γύρο των ερωτήσεων και ξεκινάμε με την κυρία Ραφάλσκα, 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κύριε κυρίες και κύριοι. Συζητάμε την κοινωνική Ευρώπη, μια ανθεκτική και ισχυρή Ευρώπη και μια δίκαιη μετάβαση. Όλα αυτά ακούγονται εξαιρετικά, αλλά απέχουμε πολύ από την υλοποίηση των στόχων αυτών. Περιμένουμε την δίκαιη μετάβαση και τα λέω αυτά ως Πολωνοί, διότι έχουμε δαμόκλειο σπάθη πάνω από το κεφάλι μας διότι ε, ε, απειλείται η Πολωνία με διακοπή της χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι κάποιοι θεωρούν ότι δεν ε, εφαρμόζεται το κράτος δικαίου. Ε, απειλούμεθα λοιπόν και η δίκαιη μετάβαση είναι όνειρο απατηλό. Μιλάμε για ψηφιακή μετάβαση και περιβαλλοντική μετάβαση. Πρόκειται λοιπόν για διτή προσέγγιση. Λέμε όμως επίσης ότι θέλουμε να διατηρήσουμε την αλληλεγγύη και θέλουμε καινοτομία και ανταγωνιστικότητα. Πώς θα τα συνδυάσετε όλα αυτά. Επίσης, όσον αφορά την ενεργειακή ένδια, είναι σημαντικό το πρόβλημα αυτό και για την Πολωνία. Το θέμα αυτό συνδέεται με την Πράσινη Συμφωνία, συνδέεται και με τις ε, οικονομίες ε, χαμηλών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Θεωρείτε ότι υπάρχει, δεν θεωρείται ότι υπάρχει κίνδυνος ε, όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα των κοινωνιών μας και όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα. Κάποιοι συνάδελφοι ανέφεραν την πρόσβαση σε στέγαση και αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα, όπως είναι και η κίνδυνη για την αγορά εργασίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Έπινγκ, παρακαλώ. Έχετε το λόγο από το ECR. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια ερώτηση προς τον Επίτροπο Ντομπρόφσκης όσον αφορά τη βιωσιμότητα Κύριε Επίτροπε, από ό,τι κατάλαβα, είσαστε θερμός υποστηρικτής της Πράσινης Συμφωνίας. Ε, είσαστε υπέρ ενό τεράστιου ε, σχεδίου ε, επενδύσεων για να μειωθούν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Ωστόσο, δεν έχουν αναφερθεί οι πυρηνικοί αντιδραστήρες και δεν αναφέρεται η πυρηνική ενέργεια. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι πολύ απλή. Ως ε, φυσικός, ε, πώς βλέπετε την πυρηνική ενέργεια ως ε, βιώσιμη λύση για την ενεργειακή μετάβαση και τους κλιματικούς στόχους της παρούσας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Περέιρα από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα σε όλους. παρά τις κοινωνικές και ε, περιβαλλοντικές ανησυχίες, δεν νομίζω ότι η νέα δέσμη ε, φέρνει νέες πολιτικές ε, στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Ούτε θα μπορέσουμε να ευθυγραμμίσουμε το στόχους βιώσιμης ανάπτυξης με την κοινωνική δικαιοσύνη. Αντιθέτως, θα αυξηθεί η εκμετάλλευση των εργαζομένων, θα έχουμε μεγαλύτερη ε, ελευθερώση και ξεπούλημα στρατηγικών τομέων. Θα πρέπει να διασφαλιστούν ε, τα κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων. Ε, και έχουμε τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων και τον πυλώνα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δεν θέλουμε όμως να επανέλθουμε στο 19ο αιώνα, θέλουμε αξιοπρεπή ζωή χωρίς να χρειάζεται να ζητιανεύουμε θα πρέπει απερίφραστα να δηλώσουμε ότι θα πρέπει να δώσουμε σαφή απάντηση. Θα αποκλείσετε από όλους τους υπολογισμούς ε, ε, το, τις δημόσιες δαπάνες ε, καθώς και επενδυτικά προγράμματα που να συγχρηματοδοτούνται από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Αυτό μπορείτε να το συνεδεύσετε ε, με μέτρα ε, για την αύξηση του εισοδήματος των, των φτωχών ή τουλάχιστον να μην εμποδίσετε τα κράτη-μέλη να το κάνουν αυτό αν το επιθυμούν. Ευχαριστώ, από την Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι πολύ ενδιαφέρον που ακούμε αυτούς που χαράσουν την πολιτική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θλίβονται για, ε, για τον περιορισμό των συλλογικών διαπραγματεύσεων και το πώς αυτό συνδέεται με την μία αύξηση μισθών ε, κλπ. Διότι στο κάτω-κάτω της γραφής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν ε, ε, ένας από τους βασικούς παράγοντες που οδήγησαν σε απορρίθμιση των αγορών. Ιδιαίτερα στη δική μου χώρα κατά τη διάρκεια της προσαρμογής που η Τρόικα ε, κυριαρχούσε. Ενδιαφέρον λοιπόν είναι που βλέπουμε αυτή τη στροφή ε, από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα ήθελα να ρωτήσω, τα εννοείται όλα αυτά στα σοβαρά. Θα το δούμε αυτά ε, όσον αφορά την Πορτογαλία και άλλε συγκρίσιμε χώρε, γιατί τα τελευταία 15 χρόνια βλέπουμε τελείω άλλα πράγματα. Η ερώτησή μου είναι η εξή πάντω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει όλο και περισσότερου ε, κοινωνικού και περιβαλλοντικού στόχου, γίνεται όλο και πιο φιλόδοξη. Και είναι πολύ ασυνήθιστη αυτή η πράσινη συμφωνία, διότι δεν ε, συνδέεται με πολλά χρήματα. Ελάχιστοι πόροι ε, αναφέρονται. Έχουμε την πολιτική συνοχή και κατόπιν αναφέρεται ένα τρισεκατομμύριο, το οποίο εμφανίστηκε από το πουθενά. Δεδομένης της πίεση ε, που ασκείται ακόμη σε χώρες όπως είναι η Πορτογαλία για δημοσιονομικό πλεόνασμα, ε, και παρά τις επιτυχίες της ε, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει να επιπλήττει τις χώρες αυτές. Από πού θα έρθουν τα χρήματα. Η κυρία Λάνιεντζ ευχαριστώ πολύ, θα μιλήσω γερμανικά. Δίδεται η δυνατότητα να ακολουθήσουμε τη διαδικασία Catch the Eye. Δύο έχουν ζητήσει το λόγο, θα τους δώσω το λόγο και κατόπιν θα προχωρήσουμε στις απαντήσεις και κατόπιν θα κλείσουμε την συζήτηση. Ο κύριος Λευτέρης Νικολάου και η Ελέν Φρίτσον. Ε, οι δύο αυτοί οι βουλευτές θα πάρουν το λόγο, ε, διότι δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ε, θα μιλήσω στα ελληνικά. Θα μιλήσω στα ελληνικά. The floor is yours. Okay. bitte. Ευχαριστώ τις εκτιμήσεις σας χαρακτηρίζει ανησυχία για νέα καπιταλιστική ύφεση και κρίση. Αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κυβερνήσεις μείωσαν μισθούς, ξεχαρβάλωσαν συλλογικές συμβάσεις, ασφαλιστικά δικαιώματα, με αφορμή την προηγούμενη κρίση, τώρα πάνω σε αυτό το έδαφος ακριβώς τρέφεστε στην ψηφιακή οικονομία, στην πράσινη ανάπτυξη. Οι προβλέψει όμω από την εφαρμογή των τεχνολογικών καινοτομιών στα πλαίσια αυτή τη καπιταλιστική οικονομία είναι δυσίωνε για του εργαζομένου, αφού φαίνεται ότι θα χαθούν χιλιάδε θέσει εργασία. Αντί αυτέ οι τεχνολογικέ καινοτομίε να ανακουφίζουν του εργαζόμενου, να βελτιώνουν τι συνθήκε εργασία. Και υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα. Η απολιγνητοποίηση απαιτεί την περιττέρω ιδιωτικοποίηση τη ΔΕΗ στην Ελλάδα. Με αποτέλεσμα 5.000 απολύσει, ένταση τη ενεργειακή φτώχεια και τη ενεργειακή εξάρτηση. Ενώ σήμερα υπάρχει τεχνολογία για καθαρότερη και αποδοτικότερη παραγωγή ενέργεια από το λιγνίτη ετοιμάζεται η εκποίηση της Λάρκο, μιας εταιρεία στρατηγικής σημασίας στον κλάδο του μετάλλου και των εξορίξεων. Αντί να ενισχυθεί η παραγωγική της ικανότητα, να επεκταθεί και σε άλλους τομείς, δημιουργώντας έτσι νέες θέσει εργασία, προετοιμάζεται για εκαθάριση, πετώντα στο δρόμο το καταρτισμένο εργατικό δυναμικό τη. Πώ τοποθετείται λοιπόν η Επιτροπή στην ανάγκη που υπάρχει... Sie nur eine Minute. Entschuldigung. Ένα λεπτό σας απομένει. Πώς τοποθετείται η Επιτροπή στην ανάγκη υπεράσπισης και εξασφάλισης θέσεων μόνιμης και σταθερής εργασίας, του δικαιώματος στη δημόσια δωρεάν κοινωνική ασφάλιση, να μην ξεπουληθεί ο ορυκτός πλούτος. Thank you. And now one minute to Madame Fritzon, and then we come to the answers of the commissioners. Thank you. Τελευταία Ευχαριστώ, θα μιλήσω σουηδικά. Είναι απολύτως απαραίτητο η ε, κλιματική μετάβαση να αντικατοπτρίζεται ε, στο ευρωπαϊκό εξάμεινο και την ετήσια ε, στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης και πιστεύω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε ακόμα πιο πέρα και να πετύχουμε μια κοινωνία δίκαιη και με ισότητα. Έχουμε την Συμφωνία του Παρισιού, του στόχους του ΟΗΕ. Θέλουμε όμως να έχουμε και δημοκρατική νομιμοποίηση. Θέλω να είμαι σαφής, να επικροτήσω ε, την σύνδεση με την εφαρμογή του πυλώνα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Για μένα ως σοσιαλδημοκράτη ε, είναι ε, αποφασιστικής σημασίας να έχουμε δίκαιη κλιματική μετάβαση που πρέπει να οικοδομείται πάνω σε ευθύνη και αλληλεγγύη με χώρες και ανθρώπους για να μην μείνει κανείς πίσω. Θα χρειαστούν συγκεκριμένα μέτρα και προσβλέπω στην συμπερίληψη του κοινωνικού ε, πυλώνα και να αυξήσουν όλα τα κράτη-μέλη τις φιλοδοξίες τους. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Δομπρόφσκης πρώτα για να απαντήσει. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Θα αρχίσω με την Πρώτη ερώτηση για τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού και την Συμφωνία. υπάρχει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, γιατί θέλουμε να, τηρού, να τηρείται το κράτος δικαίου και πρέπει να διασφαλίσουμε πράγματι ότι αυτό θα γίνεται. Εξού και σύνδεση αυτή με το κράτος δικαίου. Έπειτα. Για την ερώτησή σας για τη σύνδεση της αντικονιστικότητας της οικονομίας μας με την Πράσινη Συμφωνία και τη δίκαια μετάβαση. Μελέτες που έχουν γίνει καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θα βοηθήσει με ε, θετικές επιπτώσεις επί της οικονομίας και της απασχόλησης σε ένα βαθμό. Βέβαια, μπορεί η κατανομή να μην είναι απόλυτα ισότιμη. Κάποιες θέσεις απασχόλησης, όπως τον ανθρακορίχων για παράδειγμα, θα εξαφανιστούν. Αλλά γι' αυτό πρέπει να φροντίσουμε, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους και τις περιοχές εκείνες του κόσμου που θα πληγούν από την μετάβαση αυτή. Και έτσι έρχομαι στην άλλη ερώτηση που έγινε για τον μηχανισμό δίκαιας μετάβασης. Υπογραμμίζω πρώτα απ' όλα ότι οι χώρες μέλη τώρα πρέπει να παρουσιάσουν στρατηγικές αναπεριφέρεια δίκαιας μετάβασης για τις οποίες θα μπορέσουν να λάβουν πόρους και κονδύλια από το Ταμείο Αυτοδικαίας Μετάβασης. Μια ερώτηση επίσης έγινε για τα πυρηνικά και την ταξινόμηση των επενδύσεων. Δεν είμαι πολύ... Ξέρω από φυσική, αλλά όχι από πυρηνική φυσική. Πάντως, πράγματι, ήταν ένα επίμαχο θέμα και συζητήσεις. Αναγνωρίζετε ότι η πυρηνική ενέργεια θα παίξει το ρόλο της στην μετάβαση αυτή ως μια πηγή ενέργειας ε, χαμηλού άνθρακα. Αλλά ακόμα είναι ανοιχτό το θέμα για το ποια ακριβώ θα είναι μεταχείριση τη πυρηνική. Ευχαριστούμε. Ο κύριο Τζεντιλόνι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σίγουρα για την πράσινη αυτή μετάβαση βλέπουμε και κινδύνους και ευκαιρίες. Υπάρχει κίνδυνος για θέσεις απασχόλησης, για την ανταγωνιστικότητά μας, ναι, βέβαια. Η ιστορική εμπειρία δείχνει ότι τέτοιες μεγάλες αλλαγές πάντα ελοχεύουν τέτοιους κινδύνους. Όμως, στο τέλος μπορούμε να πετύχουμε μία καλή ισορροπία με δικαιοσύνη, αποφεύγοντας κινδύνους όπως η κλιματική αλλαγή και επίσης όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση, τελικά θα βγούμε κερδισμένοι. Και θα βγούμε κερδισμένοι εφόσον, αν μη τι άλλο, έχουμε δύο εργαλεία στη διάθεσή μας. Το ένα να είναι αυτός ο μηχανισμός της δίκαιας μετάβασης και το δεύτερο είναι ένα νέο εργαλείο προκειμένου να προστατέψουμε τις δικές μας οικονομίες και βιομηχανικούς κλάδους. Αν βρεθούμε στην πρώτη γραμμή σε διεθνές επίπεδο για να υποστηρίξουμε τις οικονομίες μας και να τις προστατέψουμε από αθέμητο ανταγωνισμό, τότε μπορούμε να τα καταφέρουμε. Γι' αυτό ε, και δουλεύουμε πάνω σε αυτόν τον μηχανισμό για την προσαρμογή σε μια οικονομία χωρίς άνθρακα. Θέλουμε να είμαστε στην ε, πρώτη γραμμή. Δεύτερον, ναι, λέτε ανακοινώνουμε κάτι χωρίς χρηματοδότηση. Μα ξέρουμε ότι η χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό δεν είναι το ποσό που θα θέλαμε πολλοί από εμά να έχουμε. Όμως υπάρχει μεγάλη δέσμευση προκειμένου ένα μεγάλο μέρος του ευρωπαϊκού προπολογισμού να αφιερωθεί στην πράσινη αυτή μετάβαση. Και η εμπειρία που έχουμε μέχρι τώρα από το σχέδιο Juncker, όπως το ονομάζουμε, δείχνει ότι υπάρχει συγκεκριμένη μόχλευση που είναι εφικτή. Και σε αυτή την περίπτωση, κατά τη γνώμη μου, η μόχλευση αυτή θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Θα έχουμε συνεπώς, πιστεύω, πόρους για να πετύχουμε αυτή τη δίκαια μετάβαση. Ευχαριστούμε κύριε Τζεντιλόνε και ο κύριο Σμιτ τώρα. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Σύντομα, η δίκαιη μετάβαση προφανώς σε μια δίκαιη Ευρώπη είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει αν πράγματι εμείς μπορούμε να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας ε, και αν παραμείνουμε ηγέτες στον κόσμο στις νέες τεχνολογίες και στον τομέα του περιβάλλοντος. Ε, πρέπει να επενδύσουμε πολλά όμως στην κατάρτιση και στην εκπαίδευση. Έτσι θα δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης. Ε, οι δίκαιες αμοιβέ επίσης. Τώρα, για τα προβλήματα ενεργειακής πενίας. η όσο φθηνότερη είναι η ενέργεια ε, έχει σχέση το πόσο φθηνότερη από την ποσότητα που καταναλώνει κανείς. Οι σωστές κατοικίες σαν παράδειγμα ε, μειώνουν το κόστος τώρα για τα κοινωνικά δικαιώματα. Εμείς θέλουμε να σεβαστούμε τον πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων και των εργασιακών δικαιωμάτων. Τα παίρνουμε αυτά πολύ σοβαρά πια. Θα παρατηρήσατε ότι και στις συστάσεις τις οποίες δίνουμε αναχώρα, εκδίδουμε αναχώρα. Σας ευχαριστώ και σας κύριε Σμιτ. Στο τέλος λοιπόν της πρώτης σειράς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας εδώ, για τις απαντήσεις σας και για τα ερωτήματα τα οποία θέσατε κι εσείς σχετικά με τις προοπτικές τις οποίες έχουμε μπροστά μας. About people with disabilities, uh, the UNCRPD, uh, ομάδα ανθρώπων οι οποίοι έχουν περιθωριοποιηθεί κοινωνικά. Υπάρχουν άνθρωποι ε, οι οποίοι πολλές φορές δεν ακούγονται στις κοινωνίες μας, δεν εκπροσωπούνται από κάποια λόμπι και ε, θα πρέπει να μην ξεχνάμε διάφορες κοινωνικές κατηγορίες όπως και τους Ρωμά. Θα συνεχίσουμε τώρα ε, για το θέμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου τον Φεβρουάριο θα συζητήσουμε τις εγγύησεις ε, για τη νεότητα, τον ελάχιστο μισθό και τα θέματα απασχόλησης. Θα ακούσουμε με ενδιαφέρον επίσης ε, και τα μηνύματα τα οποία μας έχουν στείλει ή θα μας στείλουν και τα εθνικά κοινοβουλευτικά σώματα ε, σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Σας ευχαριστώ όλους. Θα περιμένουμε να αποχωρήσουν από την αίθουσα οι συνάδελφοι από την ε, Επιτροπή Απασχόλησης και κατόπιν θα προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, διότι ήδη έχουμε καθυστερήσει.